Σήμερα θα έχουμε την ε, πρώτη σύνοδο μετά από την αποτρόπια τρομοκρατική ενέργεια η οποία έπληξε στις 22 Μαΐου το Μάντσεστερ. Δυστυχώς. Και μετά από αυτό το τραγικό γεγονός δεν σταμάτησε η τρομοκρατία να χύνει αίμα. Είχαμε το χτύπημα κατά των χριστιανών κοπτών στην Αίγυπτο και επίσης χτύπησε στην Βαγδάτη και στην Καμπούλ. Ο, ε, αυτοί οι τρομοκράτες και είχαμε και αυτού του είδους τις βάρβαρες ανθρωποκτονίες και σήμερα θα πρέπει να καταδικάσουμε αυτές τις απάνθρωπες ενέργειες, αυτή τη βία και θα πρέπει να εκφράσουμε την αλληλεγγύη μας προς τις οικογένειες των θυμάτων. Είναι αθώα τα θύματα. Δεν έκαναν τίποτα. Έχασαν τη ζωή τους λόγω αυτού του βαρβαρισμού που δυστυχώς ακόμα διέπει τον άνθρωπο και βέβαια η φωνή του Κοινοβουλίου πάντα έτσι θα ακούγεται. Να τηρήσουμε ενός λεπτού συγγύη για τα θύματα. Θα πρέπει να ανακοινώσω προς το σώμα το εξής, λέει ο Πρόεδρος. Το ότι προ προλίγο ο Πρόεδρος το να είπε ο κ. Τραμπ να αποσύρει τη χώρα του από την Συμφωνία των Παρισίων.